Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την ε, κοινή αυτή συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Μπορούμε να εγκρίνουμε, φαντάζομαι, την ημερήσια διάταξη. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Μία επιστολή από τον πρόεδρο Χόιερ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τον πρόεδρο Σούλτς και τον Υπουργό Γκραμίνια επιστολή που σας διενεμήθη μέσω email στις 3 Δεκεμβρίου. Η επιστολή αυτή μας ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διακυβερνητικής δομής ε, της του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς επίσης και μία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ξεκινήσει από τις 16 Ιανουαρίου και μετά και Προβλέπεται επίση και ένα καθορισμό για την τριετή πρώτη περίοδο της, ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, για την πολύ έγκαιρη αυτή ανταλλαγή απόψεων, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και πολύ χρήσιμη. Ξέρετε ότι ε, έχουν ολοκληρωθεί πλέον όλε οι πτυχέ διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και καταλαβαίνουμε επίσης από την επιστολή αυτή που λάβαμε ότι έχουμε πλέον μία επιτροπή επενδύσεων, έχουμε πλέον και τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο και βέβαια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήδη έχει αρχίσει να επεξεργάζεται κάποια επενδυτικά σχέδια και θα έχουμε πλέον, φαντάζομαι, ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και ένα κατεπέκτες επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα λειτουργεί πλήρως. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, να δούμε ποιε είναι οι πρώτε προκλήσει που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να δούμε επίση και πώ θα καταφέρουμε να διαρθρώσουμε μαζί σα, καθώ επίση και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έναν συνεχή διαρθρωμένο διάλογο και βέβαια με εσά που είστε ο υπεύθυνο επίτροπο, κύριε Κατάινεν. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και επίση ε, έχουμε ταχθεί θετικά υπέρ των δικών σας αιτημάτων προκειμένου να υπάρχει μία έμπρακτη επιτόπου συνεισφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αλλά θεωρώ ότι ο πρωταρχικός μας ρόλος είναι να καταφέρουμε να θεσπίσουμε και να εξασφαλίσουμε μια δημοκρατική και κοινοβουλευτική εποπτεία της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα μια εισαγωγή από τον Επίτροφο Κατάινεν και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον εισηγητή και τους αρμοδίους σκιώδεις εισηγητές. Κύριε Κατάινεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λέω κατά Κατάινεν, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που οργανώσατε τη σημερινή συζήτηση, διότι έχουμε μια σειρά ζητημάτων για τα οποία πρέπει να συνεργαστούμε. Και βεβαίω γιατί οι ευρωβουλευτές έχουν κρίσιμο ρόλο, το ώστε να μπορέσουν να περάσουν το μήνυμα στου επενδυτέ ε, και στου όλους γενικότερα, γιατί έχουν ενημερωθεί και έχουν ενημερώσει τα κράτη-μέλη και όλους τους εμπλεκομένους. Βεβαίω είναι μεγάλη πρόκληση να περάσει ένα μήνυμα για να καταλάβουν όλοι ποιε είναι οι ευκαιρίε που προσφέρονται και από την αρχή του εργομένου έτου θα αρχίσουμε μια αρκετά σημαντική πληροφοριακή εκστρατεία, ώστε να υπάρξει πλήρη ενημέρωση και συνειδητοποίηση. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αποδίδει. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με κομισιόν και με τους ευρωβουλευτές ούτως ώστε να μπορέσουν να πετύχουν αυτή την ενημέρωση συνειδητοποίηση. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ξέρετε ότι η Επιτροπή για τις Επενδύσεις θα αρχίσει να δουλεύει από αρχάς του έτους, ήδη είχε συνετρέχει το ΕΦΣΙ και έχουμε 32 project τα οποία έχουν ήδη καλυφθεί από το ΕΦΣΙ αφορούν 17 χώρες. Πρόκειται για αυτά τα 32 σχέδια, προγράμματα, έργα τα οποία αφορούν 5 δις ευρώ σαν χρηματοδότηση και πρόκειται για εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρόκειται να οδηγήσουν σε 23 ε, δις 5 δις είναι η εγγύηση για να οδηγηθούμε σε 23 δις επενδύσεις. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο επίσης συμβάλλει σε αυτή την εγγύηση και χρηματοδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει συμβάλλει στην υπογραφή 60 συμφωνιών με διάμεσες τράπεζες για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, οι οποίε είναι οι εμπορικέ τράπεζε, οι εθνικέ τράπεζε. Οπότε έχουμε 60 τέτοιε συμφωνίε μέχρι τώρα. Αυτέ οι 60 συμφωνίε αντιπροσωπεύουν 1,5 δι ευρώ. και θα οδηγήσουν σε 20 δις που θα αποτελέσει μια επένδυση που θα χρηματοδοτήσει τις ΜΜΕ. Έτσι θα έχουμε 71.000 ε, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν. Επομένω, 1,5 δις χρηματοδότηση από, την, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που θα ενισχύσουν 71.000 ΜΜΕ. 19 με 20 δις επενδύσει θα προκληθούν, οπότε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων περί τα τέλη του έτους υπολογίζεται ότι θα έχει ένα συνολικό ποσό εάν αφήσουμε τη χρηματοδότηση των SMEs και των project ότι θα φτάσει στα 50 δις όσον αφορά τις πραγματικές επενδύσεις. Οφείλω να σας αναφέρω ότι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη κατά κάποιο τρόπο το εξή. Υπάρχει ζήτηση για τέτοια χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου. Οπότε χρειάστηκε ένα τριμωχτή ο δημόσιο τομέα, αν σε πρώτη που θα γύρω σε περίπτωση έλλειψη τέτοιου ενδιαφέροντο. Οπότε φαίνεται ότι είναι κάτι το ελκυστικό η χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Αλλά φτάσαμε στο σημείο, οπότε του χρόνου θα πρέπει να κάτσουμε και να επανεξιολογήσουμε το πού θα φτάσει η χρηματοδότηση των ΜΜΕ και κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει κάποια αύξηση ανάλογα με την ε, ζήτηση. Και τα περισσότερα από αυτά τα projects, περίπου 50% αυτών, όσα έχουν καλυφθεί από χρηματοδότηση ή ενωσιακή ε, εγγύηση, αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, αποτελεσματική χρήση ενέργειας, ενεργειακή τεχνολογία, έρευνα, ανάπτυξη, ε, ψηφιακές καινοτομίες, επίσης έχουν και κάποια πρόταση για τις ε, υποδομές, σιδηρόδρομοι και αυτοκινητόδρομοι δηλαδή. Επίσης, Περισσότερα από αυτά τα project ε, αφορούν έρευνα και αναπτύξη και όπως ε, μπορείτε να φανταστείτε αν έχουμε κάνει μια καινοτομία σε οποιοδήποτε τομέα που ακόμα δεν έχει δοκιμαστεί ε, αυτό θεωρείται ως ένα project υψηλού κινδύνου. Γι' αυτό και μιλούμε για κάποια projects που αφορούν την χρηματοδότηση υπερχρηματικού κινδύνου, αλλά έχουμε και κάποιες προκλήσει να αντιμετωπίσουμε πρώτα-πρώτα. Αυτό που σας είπα για την συνειδητοποίηση, για την ενημέρωση, γιατί άπαξ και η Επιτροπή Επενδύσεων θα αρχίσει να λειτουργεί από αρχά σε επομένου έτου, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την αρχή τη προσθετικότητας. Πάρα πολύ σημαντικό όπω όλοι γνωρίζουμε και ενδεχομένω υπάρξει περιθώριο για ε, να έχουμε την ενδελεχέστερη ρύθμιση που θα μας οδηγήσει στο να δημιουργήσουν όλα τα project πως τη θέμενη αξία και για να μπορέσουν να προσθέσουν τα πράγματα η, η ΕΤΕ ε, χρηματοδοτεί 70-80 δις και το ΕΨΙ θα έρθει να συμπληρώσει αυτές τις ε, ενέργειες της ΕΤΕ. Δεν έχω τώρα τις λεπτομέρειες, τις τεχνικές για κάθε project, αλλά ίσως υπάρχουν και κάποιε οριακέ περιπτώσει όσον αφορά την εφαρμογή τη προσθετικότητα. Ας πούμε ότι δεν πληρούν τα κριτήρια για την αρχή τη προσθετικότητας, αλλά θέλω να διασφαλίσω ότι θα υπάρξει όντω εφαρμογή τη προσθετικότητα. Δεύτερη πρόκληση είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες και την ιδιωτικοτομία σε σχέση με τις πλατφόρμες των επενδύσεων. Αυτό είναι ένα όχημα επένδυσης το οποίο μπορεί να έχει χαρακτήρα θεματικό ή γεωγραφικό. Να σου πω τρία παραδείγματα για τέτοιες πλατφόρμες επενδυτικές. Στην Γαλλία έχουμε τρεις περιφέρειες που θέλουν να έχουν τέτοιες πλατφόρμες για ενεργειακή αποτελεσματικότητα και συγκεντρώνουν και καλύπτουν 40.000 κτίρια. όπως ώστε να γίνει ε, ανακαίνιση αυτών, να καλυφθούν από το ΕΦΣΙ, από ιδιώτες και από το κράτος που εμπλέκονται από εκείνο Να, πώς είναι δυνατόν ε, μια μικρή επένδυση να καλυφθεί από τις εγγύσεις ε, ή από της επενδύσεις κινδύνου. Και το τελικό αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Ότι η ενεργειακή κατανάλωση αυτών των κτίριων πρόκειται να μειωθεί πάρα πολύ. Να φτάσουμε μέχρι και στο 50%. Οπότε και ο κόσμος έτσι θα εξοικονομήσει χρήματα. Επίσης, θα έχουμε και 6.500 θέσεις από αυτό το project. Άλλο παράδειγμα πλατφόρμας ε, είναι κάτι από την Δανία. Εκεί έχουμε ένα ειδικό ταμείο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εκεί έχουμε επομένω ιδιωτικέ επενδύσει σε αυτό το όχημα. Και εκεί υπάρχει από το έξι χρηματοδότηση κινδύνου, οπότε γίνεται η επιλογή τέτοιων ε, projects για την Δανία, αλλά και τις όμορες χώρες και τις χρηματοδοτήσεις. Άλλο παράδειγμα είναι κάτι διοσυνοριακό που αφορά Γερμανία και Γαλλία. Αυτή η πλατφόρμα επίσης αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, ιδίω στι περιφέρειες, είναι ότι ευκαιρίες υπάρχουν. Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε σχετικά μικρές επενδύσεις χρησιμοποιώντας αυτή τη χρηματοδότηση κινδύνου του εύση εάν δημιουργηθεί η πλατφόρμα. Αυτό τώρα μας παραπέμπει στην τέταρτη σημαντική πρόκληση. Αυτό πώς δηλαδή θα υπάρξει ενημέρωση και συνειδητοποίηση ε, της, του συμβουλευτικού κόμβου στην Ευρώπη. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστός αυτός ο κόμβος ήδη, όμως τώρα λειτουργεί. Αυτός ο κόμβος συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη από την ΕΤΕ και από την Επιτροπή για να βοηθηθούν οι περιφέρειες, τα κρατημέλη, μέλη, οι ιδιώτες επενδυτές για να βρουν χρηματοδότηση αν δεν χρειάζεται χρηματοδότηση από την ΕΕ να υπάρξουν ε, κάποια projects και υπάρξουν κάποιες πλατφόρμες, επενδύσεις κλπ. κλπ. Ήδη τώρα βοηθούμε την Ανταλουσία στην Ισπανία και άλλες περιφέρειες. Ενδιαφέρεται η Ανταλουσία να υπάρχει τέτοια πλατφόρμα επενδυτική. Χρησιμοποιεί δηλαδή την εμπειρογνωμοσύνη μας. Οπότε αυτός ο συμβουλευτικός κόμβος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εξαρτάται από τη χρηματοδότηση της Ένωσης αλλά και όταν δεν χρειάζεται τέτοια χρηματοδότηση μπορεί να βοηθήσει να έχουμε τις πλατφόρμες και να διαρθρώσουμε το project. Τέλος, Πρόεδρε, θέλω να σας αναφέρω το εξής. Έχουμε το project port που αποτελεί κομμάτι αυτού του σχεδίου, του επενδυτικού. Έχει συμφωνήσει συμβουλή και κοινοβούλιο και ουσιαστικά αυτό είναι ένα website. Εκεί η φορείς και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να εμπλακούν και είχα πάει στη Σιγκαπούρη ξέρετε όπου συνήντησα διάφορους παράγοντες και με ρώτησαν πώς μπορούν να χρηματοδοτήσουν project τέτοια και τους είπα ακριβώς γι' αυτό και υπάρχει αυτό το website Άρα χρειάζεται να υπάρξει προβολή των καλών project, διότι τώρα η ποινική θέση στην Ευρώπη ότι είναι δύσκολο για εκείνε. Α πούμε, αν έχουμε μια τράπεζα που έχει έδρα στο Λονδίνο, δύσκολο να πάει και να βρει project ε, στην Πορτογαλία, στη Φιλανδία, στη Βουλγαρία ή σε κάποια περιφέρεια της Βουλγαρίας. Οπότε αν έχουμε αξιόλογα ε, project σε αυτό το πόρτο, το, αυτό το πόρταλ τέλος πάντων, το, την πύλη την επενδυτική, μπορούν οι αξιόλογοι επενδυτές να βρουν αξιόλογα project και να τα χρηματοδοτήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα προγράμματα θα πάρουν χρηματοδότηση από το ΕΦΣΙ, από τα διαρθρωτικά ταμεία. Χωρίς όμω και αυτό να αποκλείεται. Άρα, παρακαλώ να τα πείτε αυτά στις κυβερνήσεις σας, στις περιφέρειές σας και στους ιδιώτες επενδυτές. Και αυτό το πόρταλ, αυτή η πύλη θα αρχίσει να λειτουργεί κατά το πρώτο τρίμηνο της επομένης χρονιάς. Όμως εδώ θα βάλω μια τελεία για να μπορέσουμε να έχουμε ερωταπαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε Κατάινεν για την παρουσίαση αυτή. Καταγράφουμε προφανώς όλες αυτές τις θετικές ανησυχίες μπορούμε να πούμε που εκφράσατε ότι όντως θέλετε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου η αρχή της προσθετικότητος να διέπει πλήρως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή χρήση του. Και εμείς λοιπόν θέλουμε να συμβάλλουμε προκειμένου όντως να ισχύει αυτή η προσθετικότητα. Ας ακούσουμε τώρα πρώτα τους ηγητές. Ο κύριος Φερνάνδες έχει πρώτο το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω καταρχάς εδώ πέρα τους δύο πρόεδρους που έχουμε, καθώς επίσης και τον Επίτροπο Κατάινεν, καθώς επίσης και όλο το προσωπικό και τη γραμματεία των δύο επιτροπών. Όπως εγώ, αλλά και ο κύριος Πούλμαν, ο δεύτερος συγητής, είχαμε πει ότι έπρεπε να γίνει η συνάντηση αυτή μετά από όλη αυτή την εργασία που κάναμε τους τελευταίους μήνες και ιδίω μετά το πολύ γρήγορο αυτό χρονικό διάστημα που καταφέραμε τελικά να καταλήξουμε σε μια επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό πλέον το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να αρχίσει να αποδίδει. Πρώτο ερώτημα, η προσθετικότητα. Αυτή είναι σαφής θεωρητικά όσον αφορά το επενδυτικό σχέδιο. Δεύτερον, οι στόχοι που περιλαμβάνονται στον κανονισμό αρχίζουν και είναι ορατοί. Για παράδειγμα, ο στόχος των επενδύσεων ή ο στόχος της αύξησης απασχόλησης η προώθηση, η διαφήμιση που γίνεται στο ΕΦΣΙ επαρκεί όμως. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ουσιαστικά γνωρίζουν επαρκώ την ύπαρξη του ΕΦΣΙ. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο το ΕΦΣΙ ή τουλάχιστον κάθε κράτος μέλος να προωθήσει το ΕΦΣΙ προκειμένου οι δικαιούχοι να μπορούν να αποφεληθούν περισσότερα από αυτό. Επίσης, οι επενδυτικές πλατφόρμες είπατε ότι ήδη έχουν αρχίσει να λειτουργούν ήδη έχουν δεχθεί κάποιες επενδυτικές προτάσεις και όσον αφορά την πύλη των ευρωπαϊκών επενδυτικών έργων, το mm. περίφημο αυτό πόρταλ. Και για την περίφημη αυτή ιστοσελίδα στην οποία αναφερθήκατε και στην οποία μπορούμε να ανεβάσουμε τις επενδυτικές αυτές προτάσεις, νομίζω ότι μόνο μέσα στο 2016 το Μάρτιο θα αρχίσει να λειτουργεί αυτή η ιστοσελίδα. Για ποιο λόγο αυτή η καθυστέρηση. Ήδη από την αρχή είχαμε δει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να προωθήσει περισσότερο το εύση αυτό και να προβάλλει περισσότερο το εύση στους επενδυτές. Τελευταία ερώτηση. Αν δούμε ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και έχουμε μια κάποια θεματική συγκέντρωση στις επενδύσεις και ήδη τη βλέπουμε αυτή, ενεργειακή απόδοση για παράδειγμα. Εμείς ενδεχομένως να μην θέλουμε όμως μια τέτοια θεματική συγκέντρωση και παράλληλα μπορεί συγκέντρωση να έχουμε και σε εδαφικό επίπεδο. Πώ θα αντιμετωπίσουμε τα δύο αυτά ζητήματα. Και μία ακόμα ερώτηση. Η συμφωνία με την Κίνα. Η συμφωνία αυτή έχει τεθεί σε ισχύ, μάλλον πρόκειται να ισχύσει. Ποιε ελπίδε τρέφει ω προς αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η προστατικότητα όπως σας είπα, είναι μια αρχή που ενδεχομένω να πρέπει λίγο να προσαρμοστεί περισσότερο ή μάλλον τα κριτήριά της προκειμένου να συνάδει περισσότερο με τον κανονισμό μας. Προκειμένου δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι όντως οι εγγυήσει οι οποίες οι επενδύσεις μάλλον που χρηματοδοτούνται από τα όντως μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Δεν λέω ότι ε, τα επενδυτικά έργα τα οποία έχουμε στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν ακολουθούν τα κριτήρια αυτά. Πάντω είναι πάρα πολύ σημαντικό και με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΣΙ να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ότι όντω όλε οι επενδύσει θα επιφέρουν μια κάποια προστιθέμενη αξία. Πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Μία ακόμα πρόκληση που έχουμε είναι όντω να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο το μήνυμα προ τι ε, ενδιάμεσε τράπεζε. Τι νέε ευκαιρίε δηλαδή που μπορεί να παράσχει το ΕΦΣΥ. Ήδη 60 τράπεζε, όπω σα είπα, έχουν προσυπογράψει μια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ήδη αυτό το βήμα είναι πολύ θετικό και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ε, πολύ μεγάλα αιτήματα από διάφορου φορεί όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει προφανώς να συζητήσουμε περισσότερο με τις τράπεζες και ιδίως με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο το ΕΦΣΙ. Όσα περισσότερα απτά παραδείγματα έχουμε, τόσο πιο εύκολο είναι να προωθήσουμε το θετικό αυτό μήνυμα γύρω από το ΕΦΣΙ. Όσον αφορά τώρα τις επενδυτικές πλατφόρμες, ήδη έχουν υποβληθεί κάποιες προτάσεις αλλά στην πράξη δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν συνειδητοποιήσει τις πραγματικές ευκαιρίες που έχουμε στα πλαίσια των επενδυτικών αυτών πλατφορμών και πάλι προσπαθούμε να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τα θετικά παραδείγματα που έχουμε από τις περισσότερες αυτές τις έτσι ώστε όλο και περισσότεροι φορεί από περισσότερες χώρες να τις χρησιμοποιήσουν. Επίση, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με ορισμένε χώρες και περιφέρειες που μα έχουν πει ότι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ίδρυση τέτοιων πλατφόρμων όσον αφορά τη θεματική και δαστική συγκέντρωση. όπω ξέρετε πολύ καλά, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων λειτουργεί με βάση τη ζήτηση που υπάρχει. Μέχρι στιγμή όντω η συγκέντρωση θεματική έχει παρουσιαστεί στην έρευνα και την ανάπτυξη, την ενεργειακή απόδοση και τι ανώσιμε πηγέ ενέργεια. Αλλά προφανώ υπάρχουν και επενδυτικά έργα που έχουν να κάνουν με τι υποδομέ. Τέλο, όσον αφορά την Κίνα. Ήδη διαπραγματευόμαστε με τις αρχές της Κίνας και η αρμόδια ομάδα εργασίας έχει ήδη θεσπίσει ένα χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο μέχρι το Μάρτιο θα έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε η Κίνα να επενδύσει στις υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμή οι Κινέζοι επενδύουν σε υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγοράζουν, για παράδειγμα, ενεργειακά δίκτυα ή άλλε εγκαταστάσει. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους Κινέζους προκειμένου να μπορούν να επενδύσουν πρώτα και σε κάποιες πλατφόρμες ή σε κάποια ταμεία, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να διευρύνουν κάπως το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα έχουμε μια τέτοια σχετική συμφωνία με τους Κινέζους επενδυτές. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Μπούλμαν έχει το λόγο. Κυρίε και κύριοι, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Φερνάντες. Είναι όντω πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να λάβουμε πολύ γρήγορα κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Και όντω μεσολάβησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρί να έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρίσκεστε εδώ πέρα σήμερα προκειμένου να μα ενημερώσετε για την ενδιάμεση αυτή φάση. γιατί ακόμα δεν λειτουργούν ούτε η Επιτροπή Επενδύσεων ούτε τα εκτελεστικά όργανα. Είναι διπλή λοιπόν η ευθύνη της Κομισιόν. Κύριε Κατά, είναι στο σώμα λέμε ότι το Κοινοβούλιο ως εταίρος έχει τις εξής επιθυμίες. Ως προς την εντατικοποίηση της ε, σύμπραξης Πρώτον, αλλαγή ε, ως προς το steering board. Νομίζω ότι απεσύρθη ο πρόεδρος. Τι γίνεται λοιπόν με την ενημέρωση. Ακούστηκαν φήμες ε, στις, ε, στους διαδρόμους αλλά ε, θα ήταν καλό να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία, να υπάρχει καλύτερη αν υπήρχε καλύτερη λειτουργία του ΕΦΣΙ. Επίσης, ακούσαμε για μια ισπανική εταιρεία, η οποία μάλλον ήταν αφαιρέγγια. Υπήρχαν όμως ε, κάποιες πιστώσεις που δόθηκαν σε αυτή από το ΕΦΣΙ. Ποιο είναι το κόστος από αυτό. Έχει μείνει στα πλαίσια του ΕΦΣΙ ή είναι σε κάποια άλλα πλαίσια, κάποιου άλλου ταμείου. Επίσης, ποια είναι η, η τιμολόγηση των ε, εγγυήσεων. Γιατί μέσα στην αγορά γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ε, υπάρχει στο ε, φορολογικό επίπεδο επίσης, στο δημοσιονομικό επίπεδο επίπτωση. Τέλος, υπάρχει αυτή η διαμάχη για το ποιος θα είναι ε, ο πρώτος που θα χάσει το first loss θα είναι το FC θα είναι ε, ποιος θα είναι τελικά. Μπορείτε να μας δώσετε τέτοιες, κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Thank you. Ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Κατάιν. Ο πρόεδρος του Steering Board, ο Μάρτιν Ρέβελ, άλλαξε όντως έχει αλλάξει δουλειά, έχει περάσει σε άλλο κλάδο ε, και γι' αυτό άλλαξε και ο πρόεδρος του Διευθυντικού Συμβουλίου, του Steering Board. Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι όλα θα προχωρήσουν σωστά μόλις το ΕΦΣΙ και η Επιτροπή Επενδύσεων αρχίσει ε, στις αρχές του επόμενου έτους. Τώρα για την ισπανική εταιρεία που αναφέρατε θα είμαι μάλλον λίγο επιφυλακτικός και δεν θα δώσω πολλά ε, στοιχεία και σχόλια γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, μέσα από τη δέουσα, μέσω της δέουσας επιμέλειας κάνει τον απαραίτητο δηλαδή νομικό έλεγχο για να δουν ακριβώς ε, τι συνέβη. Και όλοι ανησυχούμε ιδιαίτερα για την κατάσταση αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας. Κατανοείται όμως ότι καταρχάς η Επιτροπή δεν έχει εμπλακεί καθόλου σε αυτή τη διαδικασία της δέουσας επιμέλειας, διότι και το όνομα της εταιρείας έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, οπότε δεν θα σχολιάσουμε πολύ την κατάσταση, δεν τη γνωρίζω και ακριβώς ή πόσο σοβαρή είναι. Τώρα, για την αποτίμηση της αξίας, της τιμής τέλος πάντων, Συνήθως αυτό δεν είναι πρόβλημα γιατί στα project του ΕΤΣΕ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, η τιμή στην αγορά είναι τόσο υψηλή που αποτελεί ε, εμπόδιο για τις επενδύσεις. Όταν όμως ε, μιλάμε για πλατφόρμες ε, μπορεί να έχουμε μεγαλύτερο θέμα γιατί μιλάμε για εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και με την αποτίμηση της τιμής των δανείων, της αξίας των δανείων. Σε κάποια κράτη-μέλη, οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες δίνουν πολύ φθηνά δάνεια λόγω της κατάστασης τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη οι τιμές είναι πολύ ψηλότερες. Συζητούμε λοιπόν με τις Εθνικές Αναπτυξιακές ε, Τράπεζες αυτή τη στιγμή για να δούμε και εσωτερικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δούμε πώς θα εξετάσουμε αυτό το θέμα. Φυσικά η λύση δεν θα είναι ε, μία για κάθε περίπτωση ε, όσον αφορά στην τιμολόγηση. Η συνεργασία με τις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες ήταν πολύ σημαντική και πάρα πολλές εξ αυτών έχουν ήδη υπογράψει πράξεις σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το ΕΤΑΕ, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως όλα αυτά γίνονται ε, περισσότερο σε επίπεδο πλατφόρμας, σε συνεργασία με τις αναπτυξιακές τράπεζες. Υπάρχουν λοιπόν προκλήσεις που ακόμη πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε όσον αφορά στην τιμολόγηση των δανείων και τη συνεργασία με τις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες, αλλά συνολικά η κατάσταση είναι σχετικά καλή και η Τράπεζα της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας ήταν πολύ ε, καλή αρρωγός. Ήταν πολύ καλές αρρωγές σε αυτό το θέμα. κύριε Πρόεδρε. Χρησιμοποίησα το χρόνο μου. Έχετε πέντε λεπτά. Απλά ε, θα ήθελα μια επερώτηση να κάνω για να μπορούμε να έχουμε μια συγκεκριμένη και με νόημα συζήτηση. Ε, μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι σε, σε θεσμικές αλλαγές ε, στο FC, το έτσι δηλαδή, αλλά και στο Steering Board, στο Διευθυντικό ε, Συμβούλιο θα είστε ε, εκ των προτέρων ε, αυτοί που θα μας ενημερώνετε για το τι αλλαγές θα γίνουν για να μην ακούμε τις φήμες, να μην πρέπει εμείς να ζητάμε τις πληροφορίες και να μας δίνετε εκ των προτέρων στοιχεία για πολιτικές ή αλλαγές ή αλλαγές προσωπικού. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με την πρακτική πλευρά της συνεργασίας μας. Ναι, γιατί όχι. Είναι η απάντηση. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Επιτροπή αλλά ε, είναι αυτοί, που επιλέγουν τα μέλη του Διευθυντικού Συμβουλίου. Αν υπάρξουν αλλαγές, ε, πολύ φυσικό είναι να ενημερώνονται οι συνομοθέτες για τις συγκεκριμένες αλλαγές. Ωραία, ευχαριστώ. άρθρο 7.3 ε, το άρθρο αυτό λέει ότι τα πρακτικά του Διευθυντικού Συμβουλίου, του Steering Committee, πρέπει να είναι δημόσια. Οπότε, ε, ε, ναι, θα πρέπει να λαμβάνουμε τις πληροφορίες, αλλά θα πρέπει και αυτή η νομική διάταξη να εφαρμόζεται πλήρως. Κυρία Τεσσεμπά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον Πρόεδρο Κατάινεν που ήρθε είναι αλήθεια ότι λείπουν τέτοιε συναντήσει και καλύτερα έτσι να έχουμε από πρώτα χαιρετήσει πληροφορίε για το πώ λειτουργεί ε, το ΕΦΣΙ, γιατί η πρώτη πρόκληση που το ΕΦΣΙ πρέπει να αντιμετωπίσει, ε, εμεί θα πρέπει σε αυτό να προσπαθήσουμε ε, ιδιαίτερα, γιατί δεν γνωρίζουν και τόσο πολύ ότι υπάρχει το πρόγραμμα Γιούγκερ και όσοι το γνωρίζουν δεν ξέρουν πώς λειτουργεί. Οπότε ε, έχουμε και τους ε, ελάσσονες παράγοντες, δηλαδή κάποιες περιφέρειες, κάποιες επιχειρήσεις και δεν ξέρουν πού θα πάνε τα σχετικά χρήματα, πώς θα υποβληθούν υποψηφιότητες των projects. Ξέρω ότι δουλεύει σκληρά πάνω σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες γιατί νομίζω ότι τελικά όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την επιτυχία των projects για πέστε μας μήπως έχετε λεπτομέρειες για το πόσα projects έχουν υποβληθεί, γιατί είπαμε για 32. Ε, επίσης έχουμε 60 με το Ταμείο Επενδύσεων. Πόσες, πόσα projects έχουν ε, υποβληθεί για να μπορούμε να καταλάβουμε πώς πάει το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων και επίσης τι αναλογία υπάρχει ε, της, ε, ε τι, τι ποσοστό υπάρχει αντιστοιχίας ε, των που γίνονται τώρα σχέση με το τι προσδοκούσε η Επιτροπή. Προχωράμε καλά, ε, προχωράμε αργά. Επίση λέγατε ότι την επόμενη χρονιά μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή στην χρηματοδότηση για το Ταμείο Επενδύσεων και την Τράπεζα Επενδύσεων. Θα υπάρξει κάποια αλλαγή, εναλλαγή. Για πέστε μα ε, ε, πάνω σε αυτό τη γνώμη σα. Προ το παρόν αυτά. Κατά Ευχαριστώ πολύ. Εάν ήμουν Ευρωβουλευτής, θα έκανα το εξή. Κάπου σε κάποια περιφέρεια θα είχα εκλεγεί και εκεί υπάρχουν μισές επιχειρήσεις και οπότε θα καθόμουν να κουβεντιάσω με κάποιες τράπεζες περιφερειακές ή εθνικές και τις ε, τοπικές τράπεζες για την ευκαιρία χρηματοδότησης των ΜΜΕ, γιατί πολλές τράπεζες δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να προχωρήσουν στην χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου. Οπότε έτσι θα έστελναν το μήνυμα στις τράπεζες. Δεύτερον, τι θα έκανα. Αν υπάρχουν κάποιοι ειδικοί τομεί όπου η περιφέρεια, οι εταιρείε της περιφέρειας ειδικεύονται. Θα έρχομαι σε επαφή με κάποιες δημόσιες αρχές, ε, ίσως με κάποιο φορέα ε, της βιομηχανίας ή των επιχειρηματιών για το κατά πόσο μπορούμε να στήσουμε μια πλατφόρμα επενδύσεων ε, ούτως ώστε ακόμα και τα μικρομεσαία projects να τύχουν χρηματοδότησης γιατί πάντοτε χρειάζεται ανάληψη δράσης έτσι συνεργασία για να υπάρξει πρωτοβουλία να υπάρξει πλατφόρμα Μπορεί να βοηθήσει επίση είπαμε, και αυτό το hub, αυτή, η διαδικτυακή πύλη συμβουλευτική. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικά θα στείλουμε αυτό το μήνυμα. Κάτι άλλο για το ίδιο θέμα. Η εκπροσώπηση της Επιτροπής στα κράτη-μέλη επίσης οργανώνει συναντήσεις εκδηλώσεις με τους εμπλεκόμενους. Μπορεί να έρθει επομένω με τους εκπροσώπους τα γραφεία της τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν μπορούσατε σε επίπεδο περιφέρειας να οργανώσετε κάποια εκδήλωση. Είναι ιδιαίτερα δραστήρια η Ισπανία σε αυτό τον τομέα, ε, αλλά και στην Γαλλία τα γραφεία της Επιτροπής ε, έχουν πει δραστηριότητα, αλλά και σε άλλες χώρες. Αυτές οι εκδηλώσεις θα μπορούσαν να στείλουν το μήνυμα στη βιομηχανία, στους επιχειρηματίες, στα ειρηνικά κέντρα, στα πανεπιστήμια. Ποσοστό επιτυχίας. Δύσκολο. Γιατί αυτοί που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων είναι κάποια project τα οποία έχουν τη χρηματοδότηση της ΕΤΕ. Άρα, εάν κάποιος θέλει χρηματοδότηση κινδύνου θα πρέπει να συμπαθεί με την ΕΤΕ είτε από τη χώρα του είτε κατευθείαν στο Λουξεμβούργο. Θα αναλυθεί το project και εάν η Τραπεζά Επενδύσεων θεωρεί ότι είναι επιλέξιμη για φυσιολογική χρηματοδότηση ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου θα σας παραπέμψει στο ΕΤΕ. Δεν ξέρω και πόσες εκατοντάδες αιτήσει έχουν ε, υποβληθεί και πόσες από αυτές θα πάνε στο Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ. Άρα, δύσκολο να καθορίσω το πόσο στο επιτυχία. Τέλος. Έκανα λάθος. τα projects δεν αφορούν 17, αλλά 13 χώρες. Και οι συμφωνίες για τις ε, ΜΜΕ είναι για 12 χώρες. Και κάποια από αυτά τα project, τα έγκριθέντα, μιλώ για τα 32, έχουν δημόσιο χαρακτήρα με την έννοια του ότι έχουν κλείσει διαπραγματεύσει, αλλού έχουν συνεχιστεί έω ότου υπογράψει ο δικαιούχο. Αλλά πάντως κάθε project τελικά θα έχει τέτοιο δημόσιο χαρακτήρα. Δηλαδή, Και έχουμε τώρα 13 τέτοια. Μπορείτε να τα βρείτε στο website της ΕΤΕ. Όλα, όλα, όλα όσα υπογραφούν θα έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Αλλά πάντως συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Thank you very Ευχαριστούμε πολύ, Ότμαν Κάρας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή τη συζήτηση τη ζητήσαμε, γιατί για μας το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει απλώς με την απόφαση. Έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον και, υπάρχει και υπάρχουν πολλές απαιτήσει από το ΕΦΣΥ. Το ΕΦΣΥ δεν είναι ε, ένα απλό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, νομίζω ότι οι πληροφορίες επίσης πρέπει σημαντικά να βελτιωθούν για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Και υπάρχουν φήμες ότι θα είναι ένα επιπλέον εργαλείο της ε, ΕΤΕΠ. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην, ε, στο home page της ε, τράπεζας έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι νομικά υποχρεωμένη να δημοσιοποιεί αυτά τα project. Οπότε ίσως υπάρχει αντίφαση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην ουσία παραβαίνει αυτή τη νομική της υποχρέωση. Δεν θέλετε να πείτε ονόματα από ό,τι καταλαβαίνω για την εταιρεία, αλλά πώς μπορεί, καλύτερο, πώς μπορεί να γίνει ώστε να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση των project και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα με εταιρείε μια εβδομάδα μόλις μετά την εξέταση, την αξιολόγηση, πώς παίρνουν τις άδειε και τελικά διακηρύσσονται αφαιρέγγες αυτές οι εταιρείε. Ε, ίσως πρέπει η αξιολόγηση που έγινε σε όλη την Ευρώπη να αλλάξει, να δούμε πώς ήταν οι επιπτώσεις της και πολλοί από εμάς βλέπουμε ότι και η τιμολόγηση των ε, εγγύσεων είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί χρησιμοποιεί το εσωτερικό ρίσκο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι απαιτήσει ε, της AB, ε, ε, ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πηγαίνουν κατευθείαν στο ΕΦΣΥ. Υπάρχουν παραδείγματα που δείχνουν ακριβώς ποια είναι η αλληλεπίδραση του ιδιωτικού κεφαλαίου και της ευθύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πώς λειτουργεί και κατά πόσο η εξέταση, αυτή η αξιολόγηση μειώνει αυτό το ρίσκο, ε, δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πιο αποδοτικά ιδιωτικά κεφάλαια. Αν το εσωτερικό ρίσκο ήταν ε, μικρότερο, τα μεγάλα project θα ήταν πιο αποτελεσματικά και αν υπήρχαν προβλήματα ε, σε αυτά δεν θα είχε πρόβλημα και η τράπεζα λόγω ε, της ε, εξάρτησής της από αυτά. Ευχαριστώ πολύ. E e. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάνει πολύ σημαντική δουλειά γιατί δημοσιοποιεί όλα τα project πριν ε, κάνει κάποια ανακοίνωση ή κάποια έκθεση αναφορά στο Κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο. Δηλαδή γίνεται δύο φορές το έτος ε, αυτή η δημοσιοποίηση, μια φορά στο Κοινοβούλιο, μια φορά στην Κομισιόν, έτσι ώστε να δει κανεί ποιε είναι οι δυνατότητε που δίνει το ΕΦΣΥ. Είναι πολύ καλό που δημοσιοποιούν λοιπόν τα project μόλι αυτά υπογραφούν. κάνουν ε, τον ευαίοντα νομικό έλεγχο όπως έκαναν και στο παρελθόν η, τράπεζα. Πρέπει όμως να είμαστε προετοιμασμένοι για απώλειες, ε, για ζημίες. Διότι ναι μεν προσπαθούμε να αποφύγουμε τις ζημίες, αλλά υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να επέλθουν ζημίες. Βέβαια είναι άλλο να έχουμε την αφηρεγγιότητα πριν ξεκινήσει το project. Αν υπάρχει λοιπόν ένα ε, έργο μεγάλου κινδύνου και μέρος του ρίσκου αυτού πραγματοποιηθεί, είναι διαφορετικό από το να χρηματοδοτήσεις μια εταιρεία η οποία είναι αφαιρέγγια ή έχει προβλήματα πριν ξεκινήσει η επένδυση. Όπως σας είπα λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσπαθεί τώρα να βρει τα γεγονότα, τα στοιχεία αυτής της συγκεκριμένης υπόθεσης και θα έχουμε περισσότερα να πούμε αργότερα για αυτό το θέμα. Το FC είναι πιο ακριβό από τη τιμή της αγοράς. Αν δούμε στην ουσία τι συμβαίνει στην αγορά. Ε, αν η αγορά ήταν πιο φθηνή από το ΕΦΣΥ δεν θα χρειαζόταν το ΕΦΣΥ γιατί θα χρηματοδοτούσε το project η αγορά. Ε, και το ΕΦΣΥ θα χρηματοδοτούσε μόνο τα project που δεν μπορούν να πάρουν χρήματα από την αγορά. Η συζήτηση τώρα για την τιμολόγηση ε, έχει γίνει μεταξύ των Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών και του ΕΦΣΥ ή της EIB. Είναι ένα τυπικό ζήτημα και όπως είπα πριν, οι όροι για την εξέβρεση κονδυλίων από την πλευρά των αναπτυξιακών τραπεζών έχει να κάνει με τα κράτη-μέλη. Η Γερμανία έχει πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και έχει πολύ χαμηλό κόστος χρηματοδότησης. Σε άλλες χώρες όμως δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα τιμολογήσουμε τον κίνδυνο και πώς θα λειτουργήσει η χρηματοδότηση. Θέλουμε να αποφύγουμε περιπτώσεις που η τιμή οι, τέλος πάντων οι εγγυήσει σπαταλώνται για πολύ ψηλές ε, τιμές και πολλές φορές όταν όλες οι τράπεζες έχουν την ίδια τιμή αυτό δεν συσχετίζεται άμεσα με την κατάσταση στην πραγματική αγορά οπότε αυτό πρέπει να το δούμε και να βρούμε μια λύση. Πραγματικά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ζημίες. Μην απογοητευτείτε αν συμβεί κάτι τέτοιο, κανείς δεν θέλει τις ζημίες, όμως αυτό είναι μέρος της πραγματικότητας ε, της ε, χρηματοδότησης υψηλού ρίσκου. Οπότε, αν τα έχουμε τρέσει σωστά, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερο το EFSI ως τώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ήταν πολύ δραστήριο όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η Βουλγαρία επίσης έχει δημιουργήσει έναν τοπικό κόμβο συμβουλευτικό σε συνεργασία με το ΕΦΣΥ για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό ε, γίνεται εδώ και κάμποσο καιρό, οπότε υπάρχουν καλά παραδείγματα κρατών μελών ή περιφερειών που έχουν ήδη ε, επωφεληθεί. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Άσουαρθ έχει το λόγο. Όχι, δεν θέλει το λόγο, μάλιστα. Σάντερλουνς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κατάινεν. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Κάναμε μια εκτεταμένη συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και στους τριμερείς διαλόγους όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ. Και είχαμε πει τελικά ότι βρέθηκαν χρήματα από τον προπολογισμό του προγράμματος ορίστας 2020. Και η απάντηση που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα είναι μην ανησυχείτε. Ο τομέας της έρευνας θα ανακτήσει τα κονδύλια του. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε ήδη κάποια στατιστικά δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν ότι όντως τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν στον τομέα της έρευνας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα ακόμα, αλλά αν δείτε την φύση των επενδύσεων θα συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει μια πτυχή έρευνας και ανάπτυξης σε όλες τις επενδύσεις δεν θα έλεγα όλες αναγκαστικά, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, στα περισσότερα επενδυτικά έργα, έχουμε μία πτυχή έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας. Εν μέρη τουλάχιστον. Επίσης, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε την κοινοτομία και την έρευνα και την ανάπτυξη. Επί του παρόντο, στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλουμε να δούμε πώ θα χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή ακόμα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή και άλλε διάβλου, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερα επενδυτικά ταμεία, ταμεία δηλαδή που θα επενδύσουν σε περισσότερα κεφάλαια κινδύνου. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε τελικά να προωθήσουμε περισσότερο τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αν ήμουν λοιπόν στη θέση σας δεν θα ανησυχούσα πάρα πολύ για το ζήτημα αυτό, συντοπιώ ποιο είναι το ζήτημα και εμένα μου απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της καινοτομίας και της έρευνας. Μέχρι στιγμής πάντως τα πράγματα δείχνουν θετικά. Τα δύο τρίτα, τα δύο τρίτα συγκεκριμένα των, των 32 αυτών επενδυτικών έργων έχουν μία πτυχή η οποία είναι, αφορά έντονα την έρευνα και την ανάπτυξη. Mr. Torvalds. Ο κύριος Τόρβαλς έχει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο διαφορετικές ερωτήσεις για... διαφορετική κατεύθυνση. Πριν από τη συζήτηση για το ΕΦΣΥ είχαμε ήδη σε πολλέ συζητήσει της ΕΚΟΝ συζητήσει για την EIB, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία συνήθως ε, σπρώχνει ε, τις ε, κανονικές χρηματοδοτήσεις από την αγορά τις παραγωνίζει και θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Υπάρχει αυτό το crowding out και στο ΕΦΣΥ. Το δεύτερο ερώτημα είναι τις προηγούμενες πρακτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνονταν χρήματα έτσι δωρεάν. Το καλό μεταξύ τώρα είναι ότι τιμολογούμε λίγο τα χρήματα που δίνουμε. Βάζουμε μια τιμή. Επί της αρχής αυτό θα λειτουργήσει σε πιο αποτελεσματική χρήση των χρημάτων ανεξάρτητα με αυτό που είπατε ε, τρίτη φορά σήμερα για το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ζημιά, πως ε, με φοβίζει διότι μας προετοιμάζεται για κάτι που δεν θα θέλαμε να δούμε. Αλλά τέλος πάντων, βλέπετε κάποια μεταστροφή προς μια πιο αποτελεσματική χρήση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το τελικά και πρέπει αυτό να συνεχίσει και σε μελλοντικά project. Ευχαριστώ. Να πω το εξής, για τέταρτη φορά. Ε, αν πρέπει να μιλήσω για ζημίες, ε, για τέταρτη φορά θα το επαναλάβω. Ελπίζω ε, να μην εκπλαγεί κανείς εδώ στο σώμα αν μετά το πρώτο έτος έρθει το εύση εδώ ενώπιόν σας και πει ότι το ποσό των ζημίας είναι κάτι τέλο πάντων. Γιατί αυτή είναι η φύση της χρηματοδότησης ε, πνευματικού κινδύνου. Δεν υπάρχουν ε, φυσικά απώλειες ζημίας το 100% ούτε και 0%. Όσο πιο πολύ διαρκέσει ένα project, ε, αν δεν είναι 5 έτη ας πούμε, αλλά είναι 6 ένα project, μπορεί να έχει επιπλέον κόστος. Και κάποιος πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό. Τέτοιου είδους θα είναι οι ζημίες. Και αυτός είναι ο λόγος που έθεσα το ζήτημα. Τώρα για την πρώτη σας ερώτηση, το crowding out. Δεν έχω ακούσει πραγματικά ε, παράπονα, καταγγελίες ότι έχει παραγωνίσει τέτοιου είδους ε, project ε, το ΕΦΣΙ. Ίσως να προκύψει στο μέλλον κάτι τέτοιο. Έχω μιλήσει για τον, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το ΕΦΣΥ και Είπαμε ότι αυτό θα είναι και ένα από τα θέματα που ενδιαφέρουν ε, το περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμένα φυσικά, διότι είναι η ουσία, η βάση της ιδέας πίσω από το ΕΦΣΥ. Το ότι δηλαδή παίρνουμε χρηματοδότηση μέσα από το ΕΦΣΥ είναι προστιθέμενη αξίμα. Πιο αποτελεσματική χρήση των χρημάτων. είναι συγκεκριμένο και αυτό παράδειγμα. Πραγματικά διαδώστε αυτό το μήνυμα, αν το ε, θέλετε. Ο συνδυασμός του ΕΦΣΥ και των διαφορετικών ταμείων για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πανέμορφος. Υπάρχουν δύο χώρες, η Ισπανία και η Μάλτα, που έχουν χρησιμοποιήσει τα διαφορετικά ταμεία ε, για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων και αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να διαδοθεί περαιτέρω είναι ένας πολύ καλός τρόπος χρήσης συνδυασμένης του ΕΨΙ και των διατροτικών ταμείων για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να είναι και μια επενδυτική πλατφόρμα που δίνει ε, κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου και κάνει και επενδύσεις σε ε, στο μετοχικό κεφάλαιο ε, που αυτό μπορεί να είναι κάτι που απαιτείται ακόμα και στις πιο ισχυρές χώρες. Ελπίζω λοιπόν ότι θα δούμε περισσότερα παραδείγματα τέτοιου είδους ε, συνδυασμού διορθωτικών ταμείων και εύση. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να μένω και την ευριανή συζήτηση που θα έχουμε για τη διαφάνεια. Πώς μπορούμε να περιορίσουμε, κάπως να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμούς που έχουμε τους θεματικούς και τους εδαφικούς. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορές από τη μία χώρα στην άλλη και από ό,τι έχω καταλάβει οι φτωχές χώρες είναι αυτές οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η δική σας η άποψη, πώς μπορείτε να διορθώσετε την κατάσταση και ξέρετε ότι στην Ιρλανδία πραγματικά ελάχιστοι γνωρίζουν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή για το επενδυτικό σχέδιο Juncker. Πάρα πολλές και διαφορετικέ συνομασίες που χρησιμοποιούμε. Νομίζω ότι πρέπει να απλοποιήσουμε εδώ πέρα κάπως τα πράγματα και να καταφέρουμε να περάσουμε ένα πιο απλό και σαφές μήνυμα προς τους πολίτες σε όλα τα κράτη-μέλη. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτύχει το εγχείρημα σε όλα τα επίπεδα. Κοιτάξτε, το επίσημο όνομα είναι επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Και έχετε δίκιο. Μολονότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανακοινώσεις Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει όλες τις ευκαιρίες ε, που εμπεριέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και θα ξεκινήσουμε μια νέα ενημερωτική εκστρατεία ήδη από τις αρχές του 2016 προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους ε, αρμόδιους φορείς. Δεν ξέρω όμως αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα και αν έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση θα μπορούσε από μόνη τη να επιτύχει σε μια τέτοια καμπάνια ενημέρωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε και τη δική σας τη βοήθεια. Ή, για να το πω διαφορετικά, είμαστε στο ίδιο πλοίο αυτή τη στιγμή. Και όσο περισσότερο διαδώσουμε το θετικό αυτό μήνυμα, όσο περισσότερο χρησιμοποιήσουμε θετικά παραδείγματα ο καθένα από, τα κράτη, από το κράτο μέλο από το οποίο προέρχεται, για να υποστηρίξουμε το εύση τόσο το καλύτερο για όλου. Εγώ χρησιμοποίησα ένα παράδειγμα από την Ιρλανδία. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, διότι ουσιαστικά έχει να κάνει με δημόσιες επενδύσεις αυτή τη φορά. Έχουμε 20 κέντρα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης που εν μέρη χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων στην Ιρλανδία. Πρόκειται για ένα σχέδιο ΣΔΙΤ και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό πώς οι δημόσιες υπηρεσίες τελικά μπορούν να αποφεληθούν από το ΕΦΣΙΝ. Και σας παραθέτω ένα πολύ απλό παράδειγμα Παραθέτοντα αυτή την περίπτωση τη Ιρλανδία. Τέτοια ακριβώ μηνύματα, τέτοια παραδείγματα θα πρέπει να προωθήσουμε και προ άλλε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιέζουμε κανένα να χρησιμοποιήσει συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα, αλλά εφόσον κάποιε περιφέρειες ή δημόσιες αρχέ αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο επενδύσεων, τόσο το καλύτερο. Όσον αφορά τώρα τον κόμβο επενδυτικών συμβουλών, και αυτός μπορεί να μα βοηθήσει στο να διαρθρώσουμε καλύτερα θετικά επενδυτικά προγράμματα και στα πλαίσια των ΣΔΙΤ έχουμε και θετικά και αρνητικά παραδείγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τωμάς έχει το λόγο. Well, I Δεν ξέρω αν οι υπηρεσίε υγείας είναι καλό παράδειγμα για σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, αλλά σε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. κάτι που το βρήκα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη ε, Κεντρική Τράπεζα του Μοντέλου. Δηλαδή τα κράτη-μέλη μπορεί να μην μπορέσουν να συμβάλλουν αρκετά σε αυτέ τι ε, επενδύσει. Τι έχει να πείτε σε αυτό που συζητήθηκε στην ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε 10, πέντε δι, είπαμε, ε, εγγύηση που θα οδηγήσουν σε 23 δις επενδύσεις. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία που αφορούν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το EIF. Τι λέτε. Επίσης, υπάρχει κάποια ισπανική εταιρεία που εμπλέκεται. Ποιο είναι το όνομα Σανταντέρ. 125 εκατομμύρια ευρώ 50 από το στρατηγικό ταμείο επενδύσεων αλλά τι θα γίνει εάν οδηγηθεί σε ζημία αυτή η κίνηση καλύπτονται από τα κέρδη άλλων projects ή από τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. Εδώ όμως μιλάμε για αυτή την πτωχεύσα εταιρεία η οποία χρηματοδότησε και τελικά ποιος πληρώνει την ύφη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που συνέκανε καλά τη δουλειά της. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι θέμα του πώς εφαρμόζονται ε, οι διατάξεις. Πότε θα μπορέσετε να με ενημερώσετε για αυτή την υπόθεση. Γιατί επανειλημμένα μας έχετε πει ότι τώρα δεν μπορείτε να πείτε τίποτα. Οπότε και εγώ συμπεραίνω ότι αφού δεν μπορείτε τώρα στο μέλλον θα μπορέσετε. Πότε όμως... I didn't say that I cannot name the Δεν είπα. Δεν μπορώ να την κατονομάσω. Όπω είπατε είναι δημοσιοποιημένο. Αν δεν μπορώ να σχολιάσω για διάφορους λόγους. και εάν θέλετε ενδελεχεί πληροφορίε μπορείτε να σα τις δώσει η ΕΤΕ. Όχι εμείς. Η Κομισιόν δεν σχετίζεται καθόλου με την υπόθεση αυτή. Και με τη χρηματοδότηση για το έτσι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί σας δώσει τις ε, πληροφορίες που θέλετε. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, πέστε μας τι θα γίνει με τη ζημία είναι 100% βέβαιο ότι πάει στο Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Άρα εξαρτάται. Ποιο έχει χρηματοδοτήσει, το ΕΦΣΙ ή η Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν μπορώ να σα πω περισσότερο όμω. Ή ακόμα είναι θέμα που πρέπει να ξεκαθαριστεί μεταξύ της Τράπεζα Επενδύσεων και της εταιρείας κάποια στιγμή. Αυτό θα ξεκαθαριστεί σίγουρα. Δεν υπάρχει εμβολία. Δεν ξέρω γίνει με αυτό το κενό επενδύσεων, γιατί αν το δείτε μακρόπνοα, εμείς ε, ειστερούμε κατά 300 δις ετησίως. Άρα, σε μια τριετία Πάμε στα 400. Η ρευστότητα στην αγορά μας οδηγεί σε χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου. Πότε πρέπει να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα βέβαια για άρα δεν είναι το κλειδί μόνο το χρήμα. Είναι το θέμα και τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Υπάρχει αυτή η τρίτη πτυχή του θέματος και αυτό πρέπει να έχει επιπτώσεις ακόμα μεγαλύτερες από το ΕΦΣΕ. Τώρα όσον αφορά τα στοιχεία. Έχουμε 23 προτάσεις. 5 δις από το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων που θα προκαλέσουν ε, πραγματικές επενδύσεις 23 δις. Και έχουμε 60 συμφωνίες μεταξύ Ταμείου Επενδύσεων και των τραπεζών που προσωπούν 1,5 δις που πρόκειται να προκαλέσει 19 με 20 δις πραγματικών ε, επενδύσεων για τις ε, ΜΜΕ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε, ο Πρόεδρος. Κύριε Σαρτουίου. Και τώρα. Να δώσουμε το λόγο σε όσους αδέλφους θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Ένα λεπτό ο καθένα για να διατυπώσετε το ερώτημά σα. Συγκεντρώστε τι ερωτήσει και απαντήστε σε όλες μαζί, αν θέλετε, κύριε την Πρόεδρε. C'est celui-ci alors qu'il faut que j'utilise Ah, mais là, c'est là, je me microphone, le Πρόεδρε. Avez-vous compris ce que je viens de dire, interprète Que euh, maintenant. Je je viens de dire έτσι κι αλλιώς οπότε τώρα να δώσουμε το λόγο σε αυτούς τους ε, συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν μια ερώτηση έχουν ένα λεπτό έκαστος και θα απαντήσει σε όλους μαζί ο κύριος Αντιπρόεδρος. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Κατάινεν, η παρουσίασή σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ιδίως το παράδειγμα που μας δώσατε από την Γαλλία για αυτά τα 40.000 κτίρια τα οποία καλύπτονται από την επενδυτική αυτή πλατφόρμα. Εμείς πριν από μερικά χρόνια στη δική μου τη χώρα καταφέραμε να λάβουμε κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και καταφέραμε προχωρώντας στην κατάλληλη ενεργειακή μόνο των κτηρίων να εξοικονομήσουμε περίπου 40-50% της τιμής ενέργειας. Πραγματικά χρειαζόμασταν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Εμεί καταφέραμε και κάναμε τη σημαντική αυτή επένδυση χωρί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι πραγματικά απαραίτητο για τέτοιε επενδύσει. Ο κύριο Μορέλη έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να επανέλθω σε ένα ζήτημα το οποίο μα αφορά ιδιαίτερα. Αναφερθήκατε στην χρηματοδοτική συνεισφορά της Κίνας που κατά άποψή μας επιφέρει και ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή συζητούμε για το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν οι Κινέζικες Αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδέουν τα δύο ζητήματα, το ΕΦΣΙ δηλαδή και το καθεστώ οικονομία τη αγορά τη Κίνα. Γιατί στα πλαίσια αυτού του ζητήματο έχουμε και κάποια προβλήματα. Μα είπατε ότι 8 με 10 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να έρθουν από την Κίνα. Στην πράξη όμω πώ θα διακυβερνήσουμε το ΕΦΣΙ στην περίπτωση αυτή. Ο κύριος Ντονάνο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, όταν θέλουμε εντό αγωγικών να πουλήσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή το επενδυτικό σχέδιο του Juncker επιτόπου, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι κάπως προβληματικά γιατί όλα είναι κάπως ασαφή ακόμα και οι ενδιάμεσες ε, τράπεζες ε, δεν κατάφεραν τελικά να αποκριθούν στα δικά μου τα ερωτήματα όσον αφορά την ίδια τη διάρθρωση και την οργάνωση της εγγύησης που παραθέτει, που μας δίνει το σχέδιο Juncker. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αποσαφηνίσουμε περισσότερο τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση, σε τι ποσό αντιστοιχεί, τι ακριβώς καλύπτει. Είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα αυτά. Και κάτι ακόμα. Ποιε είναι οι υποστηρικτικέ δομέ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αναφερθήκατε σε επενδυτικέ πλατφόρμε που μπορούν να συγκεράσουν, να συσσωρεύσουν τι διάφορε επενδυτικέ προτάσει. Στην πράξη όμω, ποιοι μπορεί να συμμετέχουν σε μια τέτοια πλατφόρμα. Οι δημόσιε, για παράδειγμα, υπηρεσίε, οι δημόσιε επιχειρήσει, τι ακριβώ θα κάνουν. Για όλα αυτά τα ερωτήματα δεν μου έχουν δοθεί απαντήσει. Θα ήθελα λοιπόν να με βοηθήσετε δυνατόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Αντιπρόεδρε για τον ευκοδομητικό διάλογο. Θα ήθελα να θέσω τα εξή δύο σημεία. Όσον αφορά στις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες, μιλήσατε για το σημαντικό ρόλο που έχουν παίξει στην εφαρμογή του έτσι και συγκεκριμένα για τη δανειοδότηση των ΜΜΕ. όμω σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίστανται αυτές οι τράπεζες και το νομοθετικό πλαίσιο για τις ε, επενδυτικές και αναπτυξιακές τράπεζες δεν είναι καλά καθορισμένο. Βλέπετε λοιπόν να έχει ζητηθεί τεχνική βοήθεια ή ας πούμε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τη δημιουργία τέτοιων εθνικών αναπτυξιακών ε, τραπεζών και σε χώρες που η χρηματοπιστωτική αγορά δεν είναι καλά αναπτυγμένη. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι κατά τη γνώμη σας όταν δεν υπάρχει μια τέτοια εθνική αναπτυξιακή τράπεζα στερεή και πώς μπορούν να πάρουν πόρους οι χώρες αυτές από τα ΕΦΣΥ. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη ε, που έχουν τέτοιες αναπτυξιακές τράπεζες και συνεισφέρουν στο ΕΦΣΥ. Έχετε δει ε, λίγο πολύ πόσο ο συνολικός ε, στόχος επενδύσεων επηρεάζεται αν θα δοθούν πάνω από 350 δις ε, χάρη στην ε, συμβολή αυτών των Εθνικών Αναπτυξιακών τραπεζών, τραπεζών για παράδειγμα. Ο κύριος Διώτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Κατάινεν, σήμερα το πρωί ή χθες αν δεν κάνω λάθος προχωρήσατε σε ένα δελτίο τύπου Σας έλεγα κύριε Αντιπρόεδρε Κατάνιν ότι σήμερα το πρωί δημοσιεύσατε ένα δελτίο τύπου με την Επίτροπο Κρέτσου όπου λέτε ότι πρόσφατα ή μάλλον στο μέλλον θα παρουσιάσετε κάποιες προτεραιότητες όσον αφορά τις επενδύσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Πόσο σύντομα θα γίνει αυτό, μπορεί να μας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα και μπορεί να μας δώσει και κάποιες ενδείξεις όσον αφορά τους βασικούς αυτούς προσανατολισμούς. Αν δεν κάνω λάθος, αναφερθήκατε πριν από λίγο στην Ισπανία και τη Μάλτα, που από κοινού δημιούργησαν μια επενδυτική πλατφόρμα. Αυτή είναι λοιπόν η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ρούμπιγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το project. Ε, υπάρχουν 400 project τα οποία θα έχουν σχεδιαστεί μέσα από τα στα πλαίσια του late tender policy. Ε, είναι δυνατό αυτό μέσω του ΕΦΣΥ, για παράδειγμα, να υπάρχει συνεργασία με τις ε, τράπεζες στην Ευρώπη, ώστε να κατονομάζονται project ε, που δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχουν αρκετά κεφάλαια είτε από την τράπεζα είτε ίδια κεφάλαια και επίσης για περιπτώσεις που δεν υπάρχει ένα business plan που να δείχνει ακριβώς πού θα είναι το ιδιωτική συνεισφορά ε, και πού όχι ε, και πώς γίνεται πολλές φορές, τι γίνεται πολλές φορές όταν αρνούνται τα, τη χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν δεν υπάρχουν ίδια κεφάλαια. Κυρία ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την αναλυτική αναφορά στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του κλίματος. Θεωρώ συγκεκριμένα ότι αυτό είναι ένα πολύ χειρό μήνυμα που ήρθε από την διάσκεψη για το κλίμα στην, στο Παρίσι γιατί πραγματικά πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε το ΕΦΣΙ για αυτό το θέμα. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με ένα θέμα που έθεσαν και άλλοι συνάδελφοι, συγκεκριμένα την ε, προστιθέμενη αξία και την προσθετικότητα που είναι σημαντική και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και το ΕΨΙ. Έχει αυτή τη βδομάδα ε, γίνει γνωστό ότι ένα ε, νοσοκομείο στο Μπέρμιχαμ χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΦΣΥ. Υπήρχε κάποιος ιδιώτης επενδυτής και ε, υπάρχει μεγάλη κριτική σε δημόσιο επίπεδο ε, γιατί είναι πολύ κακές οι υπηρεσίες, οι συνθήκες εργασίες και φαίνεται ε, ότι έδωσε 16 δις εκατομμύρια αλλά τελικά πήρε 34 εκατομμύρια και φαίνεται ε, λοιπόν ότι καλό θα είναι να υπάρχει καλύτερη διασφάλιση για το ρίσκο, ειδικά για τους ιδιώτες επενδυτές και να κερδίζουν τελικά οι πολίτες από αυτές τις επενδύσεις. Ευχαριστώ. Ο λόγος κυρία Καπέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Κατάινεν. Είπατε ήδη ότι, είπατε ήδη ότι θα έχουμε 32 project σε 13 χώρες με 5 ε, δις ε, ε, εγγυήσεων μέσα στο FC, μέσω του FC και είπατε ότι στην αρχή του επόμενου έτους θα ξεκινήσει η Επιτροπή Επενδύσεων. Χωρίς ε, να έχουμε όμως ε, ε, τελικά τα κατάλληλα όργανα, πώς θα αποφασίσουμε για τα project, θα είναι πρόταση των κρατών μελών της Κομισιόν, πώς επιλέχθηκαν αυτά τα project χωρίς να ρωτηθεί η Επιτροπή Επενδύσεων. Και επίση είπατε ότι υπάρχει αυτή η εγγύηση των 5 δι που στην ουσία θα κινητοποιήσει 23 δι. Ένα προς 15 ακούστηκε το καλοκαίρι ότι θα είναι η, η, η, η μόχλευση. Έχετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Thank you, Chair. Um... Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε που σήμερα ήρθατε να μας συναντήσετε και να μας δώσετε τόσο πληροφορίες, τόσο περισσότερες από όσες αρχικά είχαμε για αυτά τα project και για το πώς πάνε τα project, αλλά με εκπλήσει το ότι κάποιοι συνάδελφοι εδώ κατηγορούν την Επιτροπή. Τέλος πάντων λένε ότι για την ανακοίνωση για την επικοινωνία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα δεν είναι δουλειά αυτό μόνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η υπόθεση επικοινωνία. Θα πρέπει ο καθένα από εμά, ε, αν πιστεύει σε αυτό το όραμα, να, να το κάνει, ε, να, να προπάει στην επικοινωνία για να τονώσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Γιατί οι περισσότεροι οι Ευρωπαίοι ακόμα δεν έχουν ακούσει για αυτά τα project, για κάποιε πρωτοβουλίε όπω το κόσμο και πολλέ άλλε. Ούτε γνωρίζουν το ε, ταμεία στρατικών επενδύσεων, αλλά από εμά εξαρτάται το μήνυμα να φτάσει σε όσο γίνεται περισσότερους και να μπορέσουμε να κάνουμε να εμπλακούν όλο ένα και περισσότερο. Άρα δεν πρέπει μόνο να γκρινιάζουμε, πρέπει και να λάβουμε και τις ευθύνες μας. Ξέρω κύριε Επίτροπε ότι δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται με το καθένα project χωριστά, αλλά θα ήθελα να μάθω τι γίνεται με τα project που έχουν εγκριθεί στον τομέα της παιδείας, γιατί νομίζω ότι η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον, για την ανάπτυξη της οικονομίας, για το πώς θα μπορούμε να πάει η οικονομία μας. Έτσι δηλαδή να ελκύσουμε σημαντικές επενδύσεις Οπότε αν τα πάνε καλά η ε αλλά αν δεν υπάρχουν κατάλληλες δεξιότητε, δεν μπορούμε να βάλουμε σωστό δρόμο την οικονομία. Ο Πρόεδρο. Έχω και δύο σύντομε ερωτήσει. Αναφέρατε κάποια project, οπότε σκεφτούμε ότι όσον αφορά την ε, σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα είναι κάτι που αφορά τι επενδύσει ε, του δημοσίου, οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το τι θα γίνει με αυτές τις ε, επενδύσεις και τι θα γίνει και με το δημοσίο χρέας. Δεύτερη ερώτηση. Τι θα έχουμε τώρα, μία επιτάχυνση, θα έχουμε ας πούμε ε, καθυστέρηση όσον αφορά τις επενδύσεις, ε, ταυτόχρονα θα έχουμε και αύξηση των διατάξεων Ευχαριστώ πολύ. Χρειαζόμαστε πραγματικά το εύση για τη μόνωση των κτηρίων. Άμα δεν το χρειάζεστε μην το χρησιμοποιήσετε. Για κάποιο λόγο πάντως υπάρχουν τρεις γαλλικές περιφέρειες που είπαν ε, ότι ε, μπορούν ε, να κάνουν επενδύσεις χωρίς να χρησιμοποιήσουν το ταμείο αυτό. Άλλες πάλι περιφέρειες είπαν ότι χρειάζονται το ταμείο αυτό. Η Κίνα δεν μας είπε πόσα χρήματα θα επενδύσει στις ευρωπαϊκές υποδομές, πάντως ένα πράγμα είναι σαφές. Δεν πρόκειται να επενδύσουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αυτό καθεαυτό. Άρα δεν υπάρχει λόγος να επιφέρουμε αλλαγές στην διακυβερνητική δομή του ΕΦΣΥ. Δεν πρόκειται να επέμβουν καθόλου στη δομή αυτή προφανώς μπορούν να θέλουν να επενδύσουν στα πλαίσια του ΕΦΣΑ, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είπα ότι προσπαθούμε να βρούμε άλλες μεθόδους, άλλες υφιστάμενε διάβλου προκειμένου να μπορέσουν οι Κινέζοι να επενδύσουν στην Ευρώπη. Έχουν εκδηλώσει για παράδειγμα ενδιαφέρον για επενδύσει σε πλατφόρμες ε, μεταφορών, σε υποδομέ μεταφορών. Θα μπορούσαν δηλαδή να επενδύσουν στον τομέα αυτό σε διάφορε χώρε και ενδεχομένω αυτό να ενδιαφέρει ιδιαίτερα του Κινέζου επενδυτέ. Από το να αγοράζουν απλώ ενεργειακά δίκτυα σε κάποιε χώρε, θα μπορούσαν μέσω επενδυ... Ε, ε, πλατφορμών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών να επενδύσουν ταυτόχρονα σε πολλέ διαφορετικέ χώρε. Τώρα, η εγγύηση, το ποσό της εγγύησης, το νομικό καθεστώς των πλατφορμών. Δεν υπάρχει πάλι εδώ πέρα μια ενιαία λύση, εξαρτάται από τη ζήτηση κάτι το οποίο δεν έχει περάσει ακόμα στη δημόσια συζήτηση, αλλά που είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να αποφεληθούμε πλήρω από το ΕΦΣΥ και από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι να χρησιμοποιήσετε το Ευρωπαϊκό, Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών. Αν το βάλετε ακόμα και στο Google, αυτό το EIAH, θα μπορέσετε να δείτε το σημείο επαφή στη δική σας τη χώρα, έναν αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο μπορείτε να καλέσετε και να επωφεληθείτε από τον κόμβο αυτό επενδυτικών συμβουλών. Ήδη ο Ευρωπαϊκό Αυτό Κόμβο λειτουργεί. Πρόκειται για αξιωματούχου ουσιαστικά τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι οποίοι απαντούν στα τηλέφωνα αυτά και μπορούν να σα βοηθήσουν με την επενδυτική αυτή καθοδήγηση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ιδρύει επίση και νέα γραφεία σε διάφορε χώρε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν επιτόπου κάποιου επενδυτέ, εθνικέ τράπεζε τώρα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε πολλά κράτη-μέλη να θεσπίσουν τέτοιε εθνικέ συνεπτυξιακέ τράπεζε. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, αλλά ακόμα και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια τέτοια σχέδια για τη δημιουργία τέτοιων τραπεζών, αλλά και σε άλλε χώρε. Όντω, μέσω των τραπεζών αυτών μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά μπορούμε να παρέχουμε επίση και χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή μέσω του ΕΦΣΥ. Οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες δεν είναι οι μόνες βέβαια οι οποίες μπορούν να παράσχουν τέτοια χρηματοδότηση και οι πιο παραδοσιακές εμπορικές τράπεζες μπορούν σε πολλές αγορές να αποτελέσουν ενδιάμεσους. Τώρα, η συμβολή των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ανέρχεται σε 43,5 δισεκατομμύρια ευρώ αν λάβουμε συνολικά όλες τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε όμως τις επενδυτικές αυτές πλατφόρμες προκειμένου να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τους πόρους αυτούς. Οι πλατφόρμες αυτές ουσιαστικά βοηθούν τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες να διοχετεύσουν αυτή τη χρηματοδότηση όσον αφορά τα διορθωτικά ταμεία και το πώς μπορούν να συνδυαστούν με το ΕΦΣΥ και οι σχετικές κατευθυντήρες γραμμές. Ξέρετε ότι ε, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να καταρτιστούν πλήρως αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την ε, DG Regi της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήδη μπορούμε από τώρα να σας δώσουμε μια κάποια καθοδήγηση. Προσπαθούμε απλώς να καταρτήσουμε ξεκάθαρα κριτήρια για όλους. Αν όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες ε, επενδυτικέ ήδη ιδέε μπορείτε να έρθετε σε επαφή είτε με τι υπηρεσίε επενδυτικών συμβουλών είτε με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ οι δημόσιοι επενδυτέ μπορούν και αυτοί να αποφεληθούν όπω και οι ιδιώτε επενδυτέ. Αυτό εξαρτάται πάλι από τη ζήτηση. Δηλαδή, και το ΕΦΣΥ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα απογκρίνεται σε όσου θέλουν να αποτελέσουν πελάτε του. Όπως ξέρετε πολύ καλά, στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ιδιωτικά κεφάλαια, γιατί τα κράτη-μέλη Ξέρετε ότι σε πολλέ περιπτώσει δεν μπορούν να αυξήσουν πλέον τις δημόσιες δαπάνες τους. Γι' αυτό το λόγο επικεντρωνόμαστε περισσότερο στα ιδιωτικά κεφάλαια. Αλλά προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και ένας επιμερισμός του κινδύνου μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, προκειμένου να καταφέρουμε, για παράδειγμα, να βελτιώσουμε τι δημόσιε υπηρεσίε. Τώρα το ποσοστό τη μόχλευση. Και πάλι δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή έναν μέσο όρο, είμαστε πολύ νωρίς στην όλη διαδικασία. Αν όμως ε, δείτε όλα αυτά τα επενδυτικά έργα τα οποία ήδη έχουν υποβληθεί, καταλήγουμε σε ένα ποσοστό μόκλευσης το οποίο είναι σημαντικό. Εκεί βασίσαμε και τι αρχικέ μα εκτιμήσει όσον αφορά το τομέα τη παιδεία. Τρει είναι οι ευκαιρίε που παρουσιάζονται εδώ πέρα. Πρώτον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΕΦΣΥ για κάποιε εγκαταστάσει, στα πλαίσια για παράδειγμα ΣΔΙΤ, Δεύτερον, θα μπορέσετε ενδεχομένω να χρηματοδοτήσετε δραστηριότητε έρευνα και ανάπτυξη ή κάποιε καινοτομίε στον τομέα τη παιδεία για να απτυχθούν, για παράδειγμα, νέα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπω για παράδειγμα ηλεκτρονική εκμάθηση ή e learning. Έχουμε ήδη κάποια πολύ θετικά παραδείγματα σε αυτό το τομέα. Θα μπορούσαμε έτσι όντω να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ποιότητα τη παρεχόμενη παιδεία αν πραγματικά υποβληθούν αιτήματα για χρηματοδότηση τέτοιων επενδύσεων γιατί ξέρετε ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην καινοτομία, χρειάζονται και ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταφέρουν να πτύξουν την αρχική του επενδυτική ιδέα. Και η τρίτη ευκαιρία που παρουσιάζεται στον τομέα της παιδείας είναι κάτι το οποίο επί του παρόντος μας απασχολεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να καταρτήσουν το προσωπικό τους σε συγκεκριμένες δεξιότητες. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του υφιστάμενου προσωπικού. Μου έκανε εντύπωση όταν ο ιδιωτικό τομέα μα είπε ότι ε, χρειάζονται αυτού του είδου την χρηματοδότηση, χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης για την επιμόρφωση του υφιστάμενου προσωπικού. Πάντως, εφόσον αυτό υλοποιηθεί, θα είναι πολύ θετικό γιατί θα αυξήσει και την παραγωγικότητα αυτών των επιχειρήσεων και θα ενδυναμώσει βέβαια και την ανταγωνιστικότητά τους. Θα ήθελα ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή μας ανταλλαγή απόψεων. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας, αν θέλετε να συζητήσετε με μένα τα ζητήματα αυτά. Μπορούμε να συναντηθούμε επίσης και με τους διευθυντές τόσο του ΕΦΣΙ όσο και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και προφανώς ακόμα και στις συνεδριάς των πολιτικών ομάδων μπορώ να παραστώ προκειμένου να συζητήσουμε περαιτέρω τα ζητήματα αυτά και να σε ευχηθώ και καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Όντω, ε, λίγο τελευταία στιγμή σα στείλαμε την πρόσκληση αυτή. Γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε και εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία σα υπόσχομαι όμω ότι θα εκπροσωπηθεί στην επόμενη συνεδρίασή μα και θα είναι σε θέση πραγματικά να μα εξηγήσει πώ μπορούμε τελικά να καταλήξουμε, όπω είδαμε, σε συγκεκριμένα παραδείγματα, σε ζημία ή αφαιρεγγιότητα, χωρί καν έχει ξεκινήσει η επένδυση. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε συγκεκριμένα αυτή η επενδυση ειναι πολυ σημαντικο να συνειδητοποιησουμε συγκεκριμενα αυτη περιπτωση τι ακριβώ συνέβη. Ξέρετε ότι σύντομα θα εγκρίνουμε και μια συμφωνία όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και θα έχουμε και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να μπορούμε και εμείς ως κοινοβουλευτικές επιτροπές να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς το σημαντικό αυτό πρόγραμμα επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και αν σας άρεσε το 2015 ως έτος είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει